Okay, <clears throat> dear colleagues, let's start. First of all, to my right here is a new... Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ δίπλα μου έχω έναν, α, α, όχι καινούριο φίλο, έναν παλιό φίλο σε καινούρια θέση. Καλώς όρισε ο νέος α, προσωπάρτης της ε, Επιτροπής μας και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Λοιπόν, θα είναι ε, θα έχουμε την παρουσία του κύριου Κονσάλες, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ λόγω καθυστέρηση τη πτήση, προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για τη σύνδεση τη ισότητα των φύλων και των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινήσαμε στις 11 Μαΐου με μια δημόσια ακρόαση. Οπότε, εδώ στα αριστερά μου έχω τον συμπρόεδρο, τον κύριο Πιμέντα Λόπε, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ΦΑΜ Επιτροπής Γυναικών και κατά τη διάρκεια της ε, ακρόασης κάναμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις και σχόλια για το θέμα. Και τώρα θέλουμε να μπούμε σε πιο εις βάθος συζήτηση. Καταρχάς, θα ακούσουμε τις ε, δύο εισηγήτριες, την κυρία Μπιόρκ και την κυρία Φορέντσα. Ε, η μία από την Επιτροπή είναι και η άλλη από την Επιτροπή των Γυναικών. Έξι λεπτά η καθεμία θα έχουν στη διάθεσή τους. Μετά θα κάνουμε μια συζήτηση και θα καταλήξουμε βέβαια και στα συμπεράσματα. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσω το λόγο στον κύριο Λόπες, τον συμπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Στο Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά την εμπορική πολιτική. Ξέρετε πόσο ζωηρές ήταν οι συζητήσεις για ΣΥΤΑ και ΤΙΤΙΠ. Ε, Επίση όσον αφορά τη γεωργία, τα κλωστοφαντουργικά κλπ. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και στη δική μας Επιτροπή και αλλού. Πρόκειται όμως για τομεί στους οποίου οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και υφίστανται δυσμενεί διακρίσει όσον αφορά τι οικονομικέ και κοινωνικέ συνθήκες. Σημαντικό αυτό για τη σημερινή μα συζήτηση. Να καταλήξουμε πάνω σε αυτό το θέμα, σε κάποιες συστάσεις και να δώσουμε στη Λεωνόρα Φορέντζα το λόγο πρώτα-πρώτα να μας μιλήσει για έξι λεπτά. Ελεονόρα, έχεις το λόγο. Ε, όχι, τα πω εγώ. Λέει η κυρία Μπιόρκ, αν δεν έχετε πρόβλημα, όταν είχαμε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλία στην Επιτροπή Γυναικών, πρόκειψε σαφώς ότι η εμπορική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πρόσημο σε σχέση με τα δύο φύλλα. Και όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλλων εμείς θεωρήσαμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορούμε να συνεργαστούμε ε, με την κυρία Φορέντζα. Και όπως είπατε πρόεδρε, στις 11 Μαΐου είχαμε ακρόαση. Είχαμε ακρόαση από διάφορα ιδρύματα και διάφορους φορείς Οπότε και έχουμε καταλήξει ότι το εμπόριο είναι πολύ πιο σημαντικό σήμερα από ότι την εποχή της συνθήκης της Λισαβόνας. Παλιότερα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα, τώρα όμω είναι αρμοδιότητα και των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οι εμπορικέ ε, συμφωνίε δεν αφορούν μόνο του δασμού. Αφορούν κατά κύριο λόγο και άλλα πράγματα, όπω τα πρότυπα. Αυτό το είπαμε και στην συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά δηλαδή και στη συμφωνία ΤΙΣΑ για τι υπηρεσίε. Οπότε είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτέ οι συμφωνίε δεν είναι απλώ ένα σύνθημα, ένα σλόγγαν. Και ε, ακούστηκε από την Επιτροπή ότι είναι λέει λέει trade, δηλαδή στα αγγλικά μια θηλυκή συμφωνία, δηλαδή συμφωνία που να διέπεται από ισότητα. Και επομένως θα πρέπει το τι προβάλλουμε, το τι προτείνουμε για αυτές τις ε, συμφωνίες να είναι πιο δυναμικό, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και η ισότητα των δύο φύλων. Να μην προχωρούμε επομένω μόνο με τα σλόγγαν και τα συνθήματα. Οπότε για να δούμε τι θέλουμε να αναδείξουμε από όλα αυτά. Πρώτα-πρώτα ότι οι γυναίκες ε, είναι ενεργοί παράγοντες πρωτοβουλειών, ε, προτάσεων, είναι επίσης ε, εργοδότες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες το τι συνθήκες ρυθμίζονται από τις συμφωνίες για τις γυναίκες. Και μιλώ και για τον δημόσιο και για τον τομέα. Βέβαια εξαρτάται κάθε φορά, η συμφωνία αναφορά μια ε, χώρα βιομηχανική ή μια χώρα αναπτυσσόμενη. Το εμπόριο δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Το εμπόριο είναι μια πολιτική. Οπότε ο καθένας έχει τη δική του άποψη, το δικό του όραμα, τους δικούς του στόχους και ιδέες για το τι συμβαίνει ή τι θα συμβεί με κάθε εμπορική συμφωνία. Οπότε όπως και σε κάθε πολιτική θα πρέπει και η εμπορική πολιτική να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των ε, φάρμακων, στην γενική δικαιοσύνη, στην ισότητα και θα πρέπει να βοηθά η εμπορική πολιτική και στην επίτευξη των γενικότερων στόχων που έχουμε. Οπότε πολύ σωστά και ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης παριθμών 5 επισημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως αναφέρεται στο έγγραφο βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που επηρεάζουν το θεματολόγιο του εμπορίου. Κάποιες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τις γυναίκες με χαμηλές αμοιβέ και επομένως έχουμε χάσμα όσον αφορά τις αμοιβές γιατί πέραν του θέματος της καινοτομίας βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν μετέλθει και αυτό το μέσο, δηλαδή τις χαμηλές αμοιβέ προς τις γυναίκες. Κάτι που δεν το θέλουμε. Και ακούσαμε από τους εμπειρογνώμονες την ακρόαση ότι θα πρέπει να δούμε όλα τα θέματα του εμπορίου που αφορούν τα δύο φύλλα και τις γυναίκες ως ε, καταναλωτές, την πρόσβαση σε παιδεία, σε υπηρεσίες υγείας, στο νερό. Και πριν από ένα μήνα μας τόνισαν οι ότι θα πρέπει να προέξουμε πάρα πολύ τι συνέπειε τη ιδιωτικοποίηση, ιδίω όσον αφορά κάποια αγαθά όπως το νερό, αλλά και γενικότερα τον δημόσιο τομέα και τις δημόσιε συμβάσει. Όχι μόνο δηλαδή υπηρεσίε φροντίδα ε, χαμηλά εμβόμενε για τι γυναίκε. Δεν θα πρέπει να υποβαθμίζονται σε χαμηλότερες θέσεις στην ιεραρχία γενικότερα. Ε, μέχρι τώρα η αναλυσή μας βοηθήθηκε και από τους σκιώδες ηγητές, αλλά τέλος πάντων είπαμε ότι θα πρέπει τα λόγια να γίνουν έργα, θα πρέπει να δούμε μελέτες επιπτώσεων, να δούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής και να συγκρίνουμε τις καταστάσεις πριν και μετά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας. Να δούμε τι γίνεται στους τομείς που είναι πλειοψηφία οι γυναίκε να δούμε τι πρότυπα, τι στάνταρ κυριαρχούν, να φροντίσουμε τους στόχους της βιωσιμότητας, αλλά και στον δημόσιο τομέα όλα αυτά. Και η αρρωγή μέσω του εμπορίου επίσης επηρεάζει τις γυναίκες. Άρα, να συγκεράσουμε και να συνδυάσουμε όλα τα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα συζητήσαμε επομένω όλα αυτά και σε Επιτροπή Γυναικών και σε Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Πώ θα έχουμε κάποιο είδου ε, νομοθεσία δεσμευτική, πώ θα ασχίσει η αρχή τη επιμέλεια. Βέβαια, τώρα θα δώσω τη σκητάλη στην συνάδελφο Φορέντσα, αλλά να ακούσουμε και του και ηγητέ και παρακαλώ ε, να μα πείτε τη γνώμη σα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι φυσικό φαινόμενο ε, το, το εμπόριο και η εμπορική πολιτική. Δεν είναι κάτι που ξεπηγάζει σιγά σιγά, δεν είναι κάτι που διαμαγείας ε, ωφελεί όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά την υπόθεση ε, εμπόριο και να φύγουμε από τα απλά συνθήματα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εκείνη την μεριά να πηγαίνει. Και στην αυριανή εκδήλωση, αυριανή, στο αυριανό συμπόσιο, θα μιλήσει και η Ελεονόρα και θέλουν να την ακούσω και ο καθένα βλέπει το τη σκοπιά του. Η Επιτροπή Γυναικών από τη δική τη σκοπιά, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου από τη δική τη. Ε, αλλά ε, το σημαντικό είναι να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Γι' αυτό και να δούμε τις απόψεις όλων των αρμοδίων επιτροπών αλλά και στι Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλων όσων εμπλεκόμαστε σε αυτή την υπόθεση λέει η κυρία Μπιόρκ και δίνει το λόγο ο πρόεδρος την κυρία Ελεονόρα Φορέντζα σας ευχαριστώ να σας πω σύντομα συμπληρώντα την συνάδελφο Μπιόρκ έχουμε το γνωστό έγγραφο εργασίας μετά την αρχική φάση των εργασιών μας. Και να σας πω αρχικά ότι για μένα ήταν ευχαρίστης, ήταν και τιμή να συνεργαστώ με την Μαλίν Βιόρκ γιατί έτσι μας ξανήθηκαν προοπτικές όσον αφορά το θέμα της ισότητας των φίλων και όσον αφορά την νέα ερμηνεία που θέλουμε να δώσουμε στην εμπορική πολιτική, που είναι τόσο σημαντικό θέμα, όπως τα είπε και η κυρία Μπιόρκ. Και είπαμε ότι πάει και αργά ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το θέμα και αύριο το συζητήσουμε πάντως με την Επιτροπή. Για να δούμε τώρα την ουσία του έγγραφου εργασίας από πλευράς της Επιτροπής βέβαια Διεθνούς Εμπορίου Αφετηρία είναι το ότι οι εμπορικές πολιτικές για πολύ καιρό θεωρούνται ουδέτερες από πλευράς φίλων και από πλευράς του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ε, Βεβαίω και αυτό ε, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ισχύει. Ε, επίσης έχουμε την απελευθέρωση των παγκοσμίων αγορών που σίγουρα και ωφελούν όλο τον κόσμο. Αλλά δεν είναι με τίποτα αυτό ουδέτερο. Είναι λάθος. Να δούμε ομένω ποια είναι η θέση των δύο φίλων. Εκτός από τα διευθυντικά δομικά ζητήματα θα πρέπει να δίνονται υπηρεσίες και όσον αφορά την απασχόληση της υπηρεσίες, όσον αφορά την ισότητα και στο μέτωπο του εισοδήματος, αλλά και θέση της γυναίκας και ως, καταναλωτή και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οπότε τα ξαναείδαμε κατά αυτή τη θητεία με την ε, ομάδα του Gender Mainstreaming και ε, έχουμε λάβει υπόψη μας κάποιες ε, έρευνες που έχουν γίνει με τις Μαρίτσια Φοντάνα και, και άλλες και είπαμε ότι δεν είναι τα, τα πράγματα ουδέτερα. Είναι τυφλός όποιος το θεωρεί ότι αυτό ισχύει. Πάρα πολύ καιρό η Ευρώπη αγνοούσε ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις γυναίκες από τις συμφωνίες ή από τους ΛΟΑΔ και γενικότερα για τους ανθρώπους όλους. Ε, οπότε είναι προελητικό θέμα και άρα χρειάζεται να γίνει μια καινούργια πολιτική προσέγγιση. Και επί τη βάση των ερευνών που σας είπα και αφού ερμηνεύσαμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας Ε, είπαμε και στην έκθεση που είχαμε αναλάβει για την ε, ίντα που αφορούσε ε, τη συστάσεις για την περίοδο του 2010 και μετά και συμφωνήσαμε με την κυρία Μπιόρκ ότι πρέπει να επαναλάβουμε τα συμπεράσματα εκείνα και στη νέα έκθεση ότι δηλαδή τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΔ είναι αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από αυτή τη βάση θα πρέπει να κινούμεθα όταν κλείνουμε εμπορικέ συμφωνίε. Μην λαμβάνει υπόψη μόνο την αρχή του ελευθερίου εμπορίου, του δασμού κλπ. κλπ. Και έτσι με αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατεύονται. Να υπάρχουν οι σχετικέ ρήτρε που να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα Οπότε και θεωρούμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να μην είναι απλώς μια ευχή αλλά δεσμευτικό στοιχείο των συμφωνιών. Και στη δουλειά αυτή που κάναμε είπαμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε όπως το θεματολόγιο του 2030 του ΟΗΕ, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και στο σημείο 5 αναφέραμε την ισότητα των φύλων που νομίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι προς τα εκεί θα πρέπει να πάμε, να πετύχουμε αυτό το στόχο, αλλά και ότι οι εν λόγω στόχοι, όπως και οι παρθέμων 5, ε, είναι κάτι οριζόντιου εγκάρσιο χαρακτήρα, δηλαδή αφορά όλα τα άλλα σημεία. Και με αυτό το πνεύμα δουλέψαμε. Και έχουμε τώρα τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς, τη τύπ, τίζα και σέτα, αλλά έχουμε και τις εμπορικές συμφωνίες όπως αυτή με την Ιαπωνία ή την αναθεώρηση κάποιων συνθήκων, όπως τη συμφωνία με την Χιλή, που έχουν διαφοροποιημένες επιπτώσεις όσον αφορά την απασχόληση ανδρών και γυναικών. Και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες και ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ότι όλα αυτά δεν είναι ουδέτερα όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Σας, σας τα είπε μόνο η κυρία Μπιόρκο και εγώ προσαυξάνω. Χρειάζεται επομένω να γίνει μια αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξάντε και εξπόζη αυτής της συμφωνίας και να κάνουμε τέτοιου είδους αξιολόγηση και να κάνουμε ε, υποχωρητική αξιολόγηση και υποπτία. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες νέας γενιάς. Θα πρέπει έτσι να τις ερμηνεύουμε επί τη βάση όντας των φύλων και να μην... Ε, έχουμε προβλήματα και φραγμούς ε, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε από δικαστικής ε, άποψης, ούτε σε σχέση με τις ε, επενδύσεις και να δούμε τι θα γίνει με τις του δημόσιου τομέα που και αυτές θα πρέπει να διέπονται από την ισότητα και να μην έχουμε αυτές τις αρχές μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και με τις χώρες τις ανεπτυγμένες. Είπαμε ότι και το νερό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα που έχει σχέση με το εμπόριο, η προσβασιμότητα στις σχετικές υπηρεσίες αλλά και στην παιδεία επίσης υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοούμε το ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα ε, αυτά που έκανε επίσης η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να δούμε το ότι τώρα ε, η υγεία των γυναικών θίγεται θα πρέπει επομένω και εν προκειμένου με ρήτρε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα τη γυναίκα να έχει αυτοδιάθεση, να έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το ίδιο τη το σώμα. Και έχουμε τώρα τις διαπραγματεύσει με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, Ενδεχομένω ξανανοίξει το θέμα TTIP και επομένως ε, θα αλλάξει ο ρόλος των ΗΠΑ ως εμπορικού εταίρου. Θα πρέπει, οφείλει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρεσίες να βοηθούν στην ευμερία των ανθρώπων. Και όσον αφορά τους ΛΟΑΔΑ, όσον αφορά τους συνταξίχους, όσον αφορά τους μετανάστες, είναι ομάδες ε, ευάλωτες. Θα πρέπει επομένως να προστατευτεί και η υγεία και αυτών των ε, ανθρώπων και αυτό δεν είναι θέμα περιθωριακό, είναι πολύ βασικό. Ε, η προστασία των δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ανά φύλλο. Θα πρέπει να είναι ένας πυλώνας των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι παράγον, είναι στοιχείο οριζόντιο για όλες τις συμφωνίες. Θα πρέπει επομένως, ιδίως όσον αφορά το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι να προχωρούμε. Και να υπάρχουν διατάξεις δεσμευτικές και να προστατεύονται τα όσα προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Απασχόλησης. να μην έχουμε δυσμενείς διακρίσεις για την απασχόληση σε σχέση με το φύλλο, ούτε μισθολογικό χάσμα και οι διεθνείς δεσμεύσεις για το περιβάλλον επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σε αυτές τις συμβάσεις κατά προτεραιότητα με την ε, Μαλίν όλα αυτά τα λάβαμε υπόψη στο εγγραφό μας και εγκατακλείδη θέλω να σας επισημάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αποστολή της Ένωσης και ελπίζουμε ότι το έργο μας μαζί με τους σκιώδες ηγητές και τους άλλους εμπλεκομένους θα αποδώσουν κάτι το σημαντικό και θα αλλάξει ρότα η εμπορική πολιτική της Ένωσης και θα χαρακτηρίζεται από ευαισθησία προς την ισότητα των φίλων. Eh, eh. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους ε, εισηγητέ για τις παρουσιάσεις τους. Ας περάσουμε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη των Επιτροπών. Καταρχά, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδες εισηγητέ και θα αρχίσει πρώτα η κυρία Σαΐφη, σκιώδη εισηγήτρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, Φορέντσα και Μπιόρκ για τη δουλειά τους και για αυτό το έγγραφο που μας παρουσίασαν σήμερα η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί αξία Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτή την έννοια θα πρέπει και η εμπορική πολιτική να βοηθά. Το θέμα της ισότητας για το εμπόριο και την οικονομία είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγνοήσουμε. 40% των ΜΜΕ έχουν αφεντικό καμία γυναίκα. Οπότε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γυναίκα για την στρατηγική μας, την εμπορική. Επίσης, η στρατηγική εμπορία για όλους δεν καλύπτει το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Και ελπίζω ότι με την ενδιάμεση αξιολόγηση αυτό θα διορθωθεί. Στην στρατηγική επίσης θα πρέπει το θέμα της ισότητας να καλυφθεί από τις διαπραγματεύσεις για την προσαρμογή, επικαιροποίηση τέλο πάντων της συμφωνίας με την Χιλή. Χρειαζόμαστε ενημέρωση πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τις δημόσιες κρατικές υπηρεσίες, τα λέει αυτά η, ε, το έγγραφο εργασίας, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες. Είναι, εξαιρούνται από κάθε διαπραγμάτευση. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα της πλήρους διαφάνειας για τα εμπορικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρωτοπόρο ρόλο διεθνώς για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ και έχω να σας πω ότι θέλω να λάβω το λόγο για λογαριασμό της κυρίας Ματέρα που δεν μπόρεσε να παραστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για το θάρρο και για το, το ότι ήσασταν σύντομοι. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροντρίκης Πινιέρο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε, προς τις δύο συγγήτριες Φορέντσα και Μπιόρκ. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός αυτό το έγγραφο εργασίας που μας παρουσίασαν και συμφωνώ 100% με τους στόχους. Τι λέει, ότι θα πρέπει και η εμπορική πολιτική να αντιστοιχεί και να βοηθάει στην επίτευξη του στόχου της ισότητας των δύο φύλων. Όμως, για όσο χρόνο μας μένει θα ήθελα να δούμε και το πώς θα πετύχουμε με τις εμπορικές συμφωνίες να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η εμπορική πολιτική είναι ουδέτερη. Καμία πολιτική δεν είναι. Και να δούμε σε όσο χρονομασμένοι τι μέτρα θα περιλάμβουμε σε αυτές τις συμφωνίες για να ξεπεράσουμε τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων που προκύπτουν. Να δούμε τι γίνεται με ε, τις μελέτες ε, εκ των προτέρων, να κτηνογραφούνται οι χώρες, να βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε χώρα και τι επασχόληση υπάρχει για την ε, γυναίκα, τι για τον άντρα. Και επομένως να προσέξουμε περισσότερο το πώς θα πρέπει να έχουμε συγκεντρωτικά στοιχεία ανά φύλλο. Έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σωστή διάγνωση και έτσι θα μπορούσαμε να επιφέρουμε τις αναγκαίες διορθώσεις στις πολιτικές. Επίσης, θα πρέπει να γίνει ανάλυση και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Και στην Υπουργές Συμφωνία να περιλαμβάνουμε ένα κεφάλαιο το οποίο να ασχολείται με την ισότητα των φύλων. Μιλάμε για τον μισό πληθυσμό που το δικαιούται αυτό, μισό πληθυσμό της γης. Να εξετάζονται έτσι το πώς θα εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων. Οπότε έτσι να η κατά σε κάθε χώρα με την οποία θέλουμε να συνάψουμε συνθήκη. Και έτσι να πηγαίνει κανένας με μπουσουλαυτό δηλαδή στις και μπορούμε να γνωρίσουμε το ότι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ε, ε, οποιαδήποτε πολιτική κάποιου κράτους, ακόμα και πολιτική ανταγωνισμού, τόσο ώστε να υπάρχει ισότητα. Αλλά υπάρχει και κάτι παραπάνω. Είναι σημαντικό να καλύψουμε εδώ ε, και να έχουμε μαζί μας εμπειρογνώμονες για τις εμπορικές ε, συμφωνίες, τόσο ώστε το περιεχόμενο να είναι προσεκτικό, να είναι σοβαρό και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες και ειδικού. Έτσι θα αποκτήσει αυτή η υπόθεση ουσία. Αυτό περιμένει όλος ο κόσμος. Τέτοια μπορεί να γράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, την συμφωνία με την Χιλή Πρόκειται, ξέρετε, για την πρώτη χώρα που συνέπηξε με Ουρουγουάη και με Καναδά εμπορικές συμφωνίες που έχουν ένα κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Όταν κάποια αριστερή κυβέρνηση ή κάποια φιλέτερη κυβέρνηση όπως του Καναδά θεωρείται αρκετά σοβαρό να βάζει ένα τέτοιο κεφάλαιο στην εμπορική ε, συμφωνία ε, τότε πρέπει να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα ιδεολογία, είναι θέμα δικαιοσύνη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι θέμα ισότητα. Οπότε τώρα που είμαστε στη διαδικασία επικαιροποίηση τη συμφωνία με την Χιλή, τώρα που έχουμε μια ε, επίτροπο που ασχολείται με την ισότητα και το ίδιο αφορά και τον πρόεδρο της Χιλής, α, είναι γυναίκες και άρα αυτό είναι μια ευκαιρία η συμφωνία με την Χιλή να σηματοδοτήσει τη ρότα που θα πρέπει να παίρνουν οι εμπορικές συμφωνίες. Να καλύψουν την ισότητα. Και έτσι οι οφέλης από το εμπόριο να πηγαίνουν σε όσο περισσότερο κόσμο και στις γυναίκες. Θα κάνει τη διαδρομή της αυτή η έκθεση και όλοι οι συγητές έχουμε μπλακεί και εγώ και η σιώδη του ΕΛΚ και κυρίως ε, οι συγγήτριες όλοι θα συνεργαστούμε και θεωρώ και ελπίζω ότι θα βγούμε ικανοποιημένοι από αυτή την προσπάθεια. Και τελικά η υπόθεση ισότητα θα γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ροντρίγκε Φινιέρο. Όσοι βρίσκονται στην αίθουσα θα ήθελα μήπως να συνεισφέρουν κάτι στην ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Ματέρα. Μου είπε, μια που είναι υπεύθυνη για το ΕΛΚ και την Επιτροπή Γυναικών, ότι θα ήθελε να τονίσει ότι αυτές οι συμφωνίες είναι η ευκαιρία να τονωθούν οι οικονομίες και αυτό μπλέκει και τις γυναίκες επιχειρηματίες. Θα πρέπει να μελετηθεί το πώς μέσω του εμπορίου στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης μπορούμε να βοηθήσουμε στην υπόθεση της ισότητας θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταπολεμούμε τι δεμενεί διακρίσει. Η πρόσβαση στι αγορέ επίση είναι κάτι ενδιαφέρον. Η πρόσβαση απλώ των γυναικών. Χρειάζονται προγράμματα ειδικά για να βοηθήσουν και την ε, πρόσβαση σε πιστώσει, σε υποδομέ και σε αγορέ κεφαλαίων. Λέει η κυρία Ματέρα, θα πρέπει η εμπορική πολιτική να υπάρχει και να ε, γεφυρώνεται τα κενά όπου υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με τέτοιες πολιτικές θα εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των γυναικών στις εμπορικές συμφωνίες. Τα δικαιώματα, ε, τα εργασιακά, αλλά για τις γυναίκες. Να μην έχουμε δυσμενείς διακρίσεις αυτό, να είναι κάτι κομβικό για όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπεγκίν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες. Ε, Διάβασα με προσοχή το έγγραφο εργασίας. Ε, πάντοτε έχουμε επικρίνει κάποια αρνητικά των ε, εμπορικών συνθήκων ε, κάποια αρνητικά για τις γυναίκες. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι εξελίξεις έδειξαν ότι όλες οι χώρες οι αναπτυσσόμενες έχουν γνωρίσει μέσα στην εμπορία αύξηση του ΑΕΠ. Όμως υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά το φύλλο. Απαράδεκτο είναι αυτό. Γιατί έχουμε το άρθρο 8, τα των γυναικών και έχουμε επίσης και το θέμα του άρθρου 208 της συνθήκης που αφορά την ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διατάξεις σε κάθε εμπορική συμφωνία για την ισότητα. Θα πρέπει να μπουν όλες οι γυναίκες στον παραγωγικό ιστό. Αυτό σημαίνει η χειραφέτηση και αυτό θα βοηθήσει και την αύξηση των χωρών τους. Τώρα, οι παραχωρήσεις οι για τις αντισόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν σχέση με ρήτρες ε, ισότητας ε, ανδρών γυναικών. Τα είπαν οι συνεισηγήτριες ότι αν κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, έχουμε συμφωνίες. Πρόκειται για αυτές τις ρήτρε SDS. Ε, πολλές φορές ωφελούν τις ε, πολυεθνικές και όχι ε, το, το κοινωνικό κράτος που έχουμε. Και επομένως ε, τελικά φύγονται οι πιο ευάλωτοι της κοινωνίας. Δηλαδή οι γυναίκες. Ε, κατά κλείδι έχω μία πρόταση για τις συνεισηγήτριες αν γίνεται να πούμε δύο για παραπάνω όσον αφορά την εμπορική πολιτική για τις γυναίκες εδώ στην Ευρώπη, αλλά κυρίως για την συμβολή τους σε ένα πιο δίκαιο εμπόριο με λιγότερη περιθωριοποίηση και θα δούμε πώς θα αυξηθεί η συνεργασία, πώς θα αναβαθμιστεί η εταιρική σχέση μεταξύ ε, επιχειρηματιών γυναικών στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Να δούμε πώς θα γίνει αυτή την κατεύθυνση, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ, κυρία Μπεγκίν. Η κυρία Μπιλμπάου έχει το λόγο. Ευχαριστούμε τις εισηγήτριες και τις χιώδες εισηγήτριες για όσα έκαναν. Και η δική μας πολιτική ομάδα θεωρεί ότι είναι θετικά όλα αυτά ως ιδέες. Ε, βέβαια και θα πρέπει οι διεθνεί εμπορικέ συνθήκε να βοηθούν την, εμπορική, την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση του να στρέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση της ε, συμφωνίας τρίτης γενεάς να μπορέσουμε να τους βάζουμε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο εκεί που να καλύπτονται τα δικαιώματα των γυναικών ή τέλος πάντων το πώς να ε, ξεκινούν προγράμματα για την απασχόληση των γυναικών. Γι' αυτό και συμφωνούμε όσον αφορά το να κάνουμε κάποιες μελέτες για τις επιπτώσεις των συμφωνιών αυτών και κάποιες συμφωνίες με τρίτες χώρες όπου να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούμε να δούμε πώς θα ωφελούνται από πολλές απασχόλησεις οι γυναίκες. Οπότε από αυτή την πλευρά θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν φέρει ανάπτυξη, αλλά αναφέρουν για τις γυναίκες, στη συμφωνία με κάποιες τρίτες χώρες. Να τις βελτιώσουμε και να φτάσουμε στην ισότητα. Όχι μόνο για τις χώρες με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες, να αναλυθούν οι επιπτώσεις των συμφωνιών αυτών από πλευράς απασχόλησης στις χώρες της Ένωσης. Γιατί κουράμε το δάχτυλο στις άλλες χώρες, αλλά δεν φροντίζουμε τα του οίκου μας. Δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας από πλευρά ισότητας ακόμα. Άρα έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Να λάβουμε υπόψη τις ιδιορυθμίες κάθε χώρας, αλλά να δούμε ας πούμε τι στοιχεία υπάρχουν στη για να απασχόληση των γυναικών σε κάποιους τομείς όπου ασχολούνται οι γυναίκες. Ε, σε κάποιους τομείς ε, οι γυναίκες έχουν προχωρήσει στη χειλή πολύ περισσότερο από όσο στην Ευρώπη. Άρα ανάλυση των επιπτώσεων ε, να έχουμε τα στοιχεία που αφορούν τις γυναίκες και έτσι συνολικά να πάμε προς την ισότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Λάνια. Κλείνουμε λοιπόν έτσι τη συζήτηση με τα μέλη και να ακούσουμε τώρα την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόμας Μπέρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε στη σημερινή συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πραγματικά χαιρόμαστε που μπορούμε να συμβάλλουμε. Μάλιστα είμαστε και κομμάτι της συζήτησης γιατί και εμείς αύριο οργανώνουμε ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Γυναίκες και το ε, ε, Εμπόριο μια συζήτηση με την Επίτροπο και τον κύριο Γκονζάλες. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα και θέλω να τονίσω κάποια από αυτά. Ε, τέσσερα. Σε τέσσερα θα επικεντρωθώ. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι κάνουμε σήμερα, τι δεν κάνουμε σήμερα και τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε αύριο. Θα ξεκινήσω με κάτι που άκουσα από την τελευταία παρέμβαση. Ε, η ομιλήτρια μίλησε, η ε, μίλησε λέγοντας ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό ακόμη που μπορούμε να προωθήσουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όντως μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν ξέρουμε ακόμα πολλά εξακολουθούμε να αξιολογούμε τις ε, συμφωνίες αυτές ε, και σε όλα τα στις αξιολογήσεις κινδύνου, στις αξιολογήσεις εκπός που κάνουμε, αλλά βεβαίως ε, είναι μεγάλη η πρόκληση γιατί δεν μελετούμε μόνο συγκεκριμένα δεδομένα, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το επίπεδο των δεδομένων και να δούμε θέματα ας πούμε ιδιοκτησίας, σε ποιον ανήκουν αυτές οι επιχειρήσεις, ποιος τις διαχειρίζεται. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη δουλειά και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το σημείο αυτό και το ανέφερε και η κυρία Πινιέρο ότι όντω χρειάζεται να κάνουμε μια καλή διάγνωση, μια απεικόνηση των, ε, της κατάστασης για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματά μας. Οπότε, όταν διαβάζω το, το σχέδιο έκθεσης, που έχει υποβληθεί προ μελέτη στην Επιτροπή σα, Είναι προφανέ ότι δεν είναι ουδέτερο προ το φύλλο το ε, εμπόριο. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε διάφορε υποθέσει από αυτού, αλλά στα πλαίσια μια πολιτική που βασίζεται σε αποδείξει, όντω πρέπει να μάθουμε περισσότερα και να έχουμε πρώτα τα γεγονότα πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε πολιτικέ. Πολλέ από αυτέ τι πολιτικέ και τι σχετικέ δράσει ήδη υπάρχουν, Πρόεδρε. Τώρα, τι κάνουμε σήμερα, ήδη πέραν το ότι βάζουμε το θέμα αυτό στι αξιολογήσει μα, έχουμε συγκεκριμένε δεσμεύσει αναλάβει, α πούμε, για την εφαρμογή των συμβάσεων του ILO, ε, ο στόχο τη ε, μη διακριτική μεταχείριση στην απασχόληση, ίση ε, αμοιβή. Όλα αυτά είναι απαιτήσει και για του δικαιούχου του προγράμματο gsp sin Επίση, ήδη και πολλέ φορέ σε συνεργασία με τον ΩΣΑ, και το ITC, το Διεθνέ ε, Κέντρο Εμπόριου, ασχολούμαστε με θέματα που έχουν ε, και μια πτυχή του φύλου. Οπότε κάνουμε αρκετά πράγματα ήδη σήμερα. Υπάρχουν βεβαίως πράγματα που δεν κάνουμε ακόμη. Υπάρχουν ε, κάποιες αναφορές και εντός της έκθεσης για τις ιδιωτικοποίησεις. Οι εμπορικέ συμφωνίε δεν ιδιωτικοποιούν τομεί ή υπηρεσίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει σε όλε τι στις συμφωνίες της μια ρήτρα που, τις, που μπορεί να, να εισάγει κάποιους συγκεκριμένου κανόνες όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση ενός συγκεκριμένου κλάδου. Δεν κάνουμε λοιπόν ιδιωτικοποίησεις μέσω των συμφωνιών. Και άκουσα από τα σχόλια, αλλά διάβασα και από τις εισηγήσεις, ότι υπάρχει πεδίο να μελετήσουμε κάποιε δεσμεύσει ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά για κάποιου συγκεκριμένου τομεί που είναι σημαντικοί για το φύλλο γενικώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό σημείο και πρέπει να το δούμε πιο στενά. Άκουσα από τους εμπειρογνώμονες και στην ε, ακρόαση τη 11 η Μαΐου να λένε ότι στον, ε, στις υπηρεσίες υγείας πολλές γυναίκες, ε, πολύ περισσότερο είναι το γυναικείο εργασιακό δυναμικό και εκεί μπορούν να υπάρχουν όντως ε, πολλές ευκαιρίες αν απελευθερώσουμε το δυναμικό του τομέα αυτού. Έχουμε λοιπόν ότι μεγάλο δυναμικό, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε και το άνοιγμα των τομέων που ίσως είναι λίγο πιο κλειστή σε ό,τι αφορά την ένταξή του στις εμπορικές μας συμφωνίες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που δεν κάνουμε, αλλά βεβαίω υπάρχουν και πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίω θα το συζητήσουμε και αύριο. Δεν μπορώ σήμερα ε, να σας πω, κυρία Σαΐφη, αν ε, τι θα γίνει μάλλον με τι ε, διαπραγματεύσει με τη Χιλή. Ακόμα πρέπει να υιοθετηθεί η θέση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την διαπραγματευτική εντολή. Αλλά είναι σαφέ ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα γιατί, ε, όπω είπε η κυρία Βιόρκ, πρέπει να αφήσουμε τα συνθήματα. Αλλά ε, το εμπόριο σημαίνει εμπόριο για όλου και πρέπει βεβαίω όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν και να υποφελούνται. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά το φύλλο και να μπορούμε να μελετούμε τι πολιτικέ μα σχετικά με το εμπόριο ως προς αυτή την πτυχή. Έχοντας συγκεκριμένε διατάξεις που θα φορούν τα φύλλα στις εμπορικές μας συμφωνίες. Ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω και ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί στα πλαίσια της εκθεσής σας είναι το εξή. Η, πολιτική του, η εμπορική πολιτική έχει να κάνει με την προώθηση των αξιών και των προτύπων μας στον κόσμο. Είναι δύσκολο όμως αυτό να το κάνεις όταν, ε, ε, προς τα έξω, όταν δεν υπάρχουν προς τα μέσα. Έχουμε βεβαίως υψηλά πρότυπα για διάφορους τομείς, αλλά κάποιες από τις ιδέες που ακούω και διαβάζω συμπεριλαμβανομένου και του περιορισμού α πούμε, κάποιων ρητρών για τι δημόσιε προμήθειε για συγκεκριμένε εταιρείε ή να μην του επιτρέπουμε να πάμε σε εταιρείε που αποτελούνται από αμυγό ανδρικά διοικητικά συμβούλια. Αυτά μπορούμε να τα ρυθμίσουμε στην εσωτερική μα αγορά. Αν δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε στην εσωτερική μα αγορά, δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τέτοια πρότυπα προ τα έξω. Οπότε είναι, είναι σημαντικό να έχουμε εσωτερικά καλώ εδρεωμένη πολιτική εμπορική για να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτά τα πρότυπα που έχουμε στην, στο ιστορικό της Ένωσης, να τα προωθήσουμε προς τα έξω και, και στις εμπορικές μας πολιτικές και συμφωνίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η έμπνευση που ψάχνουμε όταν θα μελετήσουμε περαιτέρω το τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής για να καλύψουμε το θέμα των φύλων. Βεβαίω, ε, με χαρά περιμένουμε την περαιτέρω συζήτηση μαζί σα και φυσικά το θέμα αυτό θα συζητηθεί και αύριο στο Διεθνέ Φόρουμ και ελπίζω πολύ να είσαστε εκεί. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και για να ολοκληρώσουμε θα δώσω το λόγο στις συζήτριες. Δεν ξέρω ποια από σας θα ήθελε να αρχίσει. Α, με την ίδια σειρά. Παρακαλώ. Η Ελεονόρα μπορεί να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ε, σκιώδεις Υπάρχει, βλέπω, μεγάλο επίπεδο δέσμευσης και πολύ εμπειρογνωμοσύνη. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ε, το έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο εργασία και όταν θα... Ε, προχωρήσουμε, θα θέσουμε και στόχους, διότι πολλοί λένε πως πρέπει να δείξουμε πως ε, το εμπόριο πρέπει να είναι για όλους και οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου νέας γενιάς πρέπει να δουν ε, όλες τις επιτυχίες. Ε, να περιμένουμε επίσης και για την εκτίμηση αντικτύπου και να πω ότι συμφωνώ με αυτά που άκουσα ότι δηλαδή πρέπει οι προτάσεις μας να είναι πιο συγκεκριμένες έτσι ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να τις υλοποιήσει. Πιστεύω πως είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν συνέπειες ε, που προκύπτουν από τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Βορρά και Νότου, μεταξύ διαφόρων τύπων οικονομίας. Ε, στην ε, περίπτωση της ΣΥΤΑ ή της ΤΙΤΙΠ, των βόρειων συμφωνιών, διαφέρουν κάπως από τις υπόλοιπες. Όμως οι γυναίκες πρέπει να ε, τις βλέπουμε ως ε, εργαζόμενες και να βελτιώσουμε ε, σημαντικά το επίπεδο των ε, υπηρεσιών και των συνθήκων. Επίσης, όπως είπε και η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να δούμε και τις δομές περί ευθύνης. Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το έγγραφο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο έκθεσης φέτος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σας πω ότι θα συνεδριάσουμε στις 22 Ιουνίου, 11 με 1 το πρωί. Θα σας στείλω και email σχετικά. Θα συνεδριάσουμε λοιπόν οι σκιώδεις συζητητές, αλλά και όχι μόνο. Θα καλέσουμε διάφορους εκπροσώπους με κυβερνικών οργανώσεων, Business Europe, ε, Oxfam και διάφορους άλλους φορείς, οι οποίοι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην έκθεσή μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, να πω καταρχάς ότι χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, όμως στην αρχή Είπατε πως δεν είστε σίγουροι για το αν υπάρχουν ε, συνέπειες ε, που αφορούν τις γυναίκες στην εμπορική πολιτική. Και εμείς θέλουμε να σας πείσουμε ε, για το αντίθετο. Προσπαθείτε μάλλον εσείς να μας πείσετε ότι δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν υπάρχει διάσταση του φίλου στις εμπορικές συμφωνίες, όμως εμείς ε, διαφωνούμε και θα συνεχίσουμε την ε, μάχη έτσι ώστε να μπορούν να το δουν όλοι. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές αναγκαστήκαμε να κάνουμε δύσκολα πράγματα, ε, ασχοληθήκαμε με εκθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα ε, των εργαζομένων, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το έργο. Ελπίζω λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας συνοδεύσει σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω όλους ε, αύριο και οι συναδελφοί μου θα είναι εδώ, η Φλωρέντσα. Ελπίζω λοιπόν ε, τα αποτελέσματα των εργασιών μας να φτάσουν και στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φορέντσα έχει το λόγο. Ε, βέβαια. Και συμφωνώ με αυτά στα οποία προβλέπει και η Μάλιν. Είμαστε αποφασισμένες να προωθήσουμε αυτή μας την ε, πολιτική προσπάθεια ούτως ώστε να είναι ευαίσθητη στο θέμα εσόδος δύο η πολιτική και η πολιτική της ε, ε, Επιτροπής γενικότερα. Ε, οπότε και εγώ συμφωνώ με τη διαπίστωσή της ε, για το ότι θα πρέπει να δούμε και αύριο τι θα διατυπωθεί στη συνάντηση της Επιτροπής των Γυναικών. Ε, ευχαριστώ τους που έλαβαν το λόγο στην Επιτροπή και επίση θα πρέπει σε αυτή την έκθεση να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι από τις δύο συναρμόδιες επιτροπές, τις επιτροπές αυτές που θα γνωμοδοτήσουν Επομένω θα πρέπει το σύντομο δυνατών να ολοκληρώσουμε την ε, έκθεση και με την άποψη κάποιων ε, ειδικών ε, και όσων ανδρών και γυναικών εμπλέκονται στην υπόθεση της σύναψης εμπορικών συμφωνιών. Επίσης σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και ιδίω για κάποια ζητήματα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτά που επισημάνατε και με την ε, κυρία Μπεγκίν συμφωνώ ότι θα πρέπει εις βάθος και περισσότερο να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των συμφωνιών για τις ε, επιχειρήσεις των γυναικών και έτσι οι γυναίκες επιχειρηματίες θα πρέπει να προτείνουν λύσεις και ιδέες για τις εμπορικές συμφωνίες που θα πρέπει ως συμφωνίες και αυτές να περιέχουν πνεύμα ευαίσθητο στον ρωτησότητα των δύο φίλων. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία του κάθε κλάδου. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιδεολογική προσέγγιση. Περισσότερη ευημερία, περισσότερη, περισσότερο ισότητα τελικά μεταξύ των δύο γυναικών. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Θα πρέπει να δούμε περισσότερο τους στόχους που έχουμε, ότι δηλαδή τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά θα πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα στις εμπορικές συμφωνίες. Άρα θα πρέπει να έχουμε και μελέτες επιπτώσεων και αξιολογήσεις. Και όπως είπε και η Μελίν, αυτό θα πρέπει να υπόψη όταν στις 27 ε, με μία συνδεθούμε με τις σκιώδεις ε, εισηγήτριες. Αυτός ο διάλογος των δύο επιτροπών για αυτή την έκθεση θα αποκτήσει περισσότερο ειδικό βάρος. Αυτή η ομάδα του mainstream θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αρχίσει μια Πάγιο χαρακτήρα συνεργασία με την Επιστροπή, το Γυναικών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και τον Αντιπρόεδρό μου. Σύμφωνα με το προσωπικό μας χρονοδιάγραμμα, η επόμενη κοινή συνεδρίαση θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου. Και νομίζω πως μετά θα έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης έτοιμο, ένα σχέδιο, ένα τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διακόψουμε τώρα για δύο λεπτά και θα συνεχίσουμε στις 4 με τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ.